Στη στρατηγική διεύνηση έχουμε μια αιτιολόγηση ψήφου από τον κύριο Πρέντα. Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ απλά να υπογραμμίσω την ποιότητα της προσπάθειας ε, του κύριου Αλμπερτίνη. Να προσθέσω επίσης ότι εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης γιατί θεωρώ ότι η διεύρυνση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Να διευκρινίσω επίσης ότι ψήφισα διαφορετικά από την πολιτική μου ομάδα σε πολλούς τομείς που έχουν σχέση περισσότερο με το κοσυφοπαίδιο και αυτό γιατί έχω μια διαφορετική άποψη από την πλειοψηφία των περισσότερων χωρών για το κοσυφοπαίδιο. Και γι' αυτό ακριβώς ακολούθησα διαφορετική στάση. Σχετικά με την τροπολογία 17 του άρθρου 19 και την τροπολογία 22 όπως και 24 και μετά από την αιτιολογική σκέψη 4 παραμένω πάντα πιστό στη θέση μου ότι η διεύρυνση είναι πολύ σημαντικό πράγμα αλλά οι διαφορές τις οποίες ε, έχουν διαφορετικές θέσεις πέντε χωρών μελών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αν θέλετε να κάνετε πηγαδάκια να βγείτε έξω από την αίθουσα. Θέλω ησυχία, παρακαλώ. Η επόμενη επεξήγηση από την κυρία Μπούρη Ρακκρίζα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ισπανική Σοσιαλιστική Αντιπροσωπεία σε σχέση με το Κόσοβο θέλουν να τονίζουν το γεγονό ότι δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς το κοσυφοπαίδιο σαν εξάρτητο κράτος. Υπήρξε μια μονομερής διακήρυξη ανεξαρτησία και μόνο από την πλευρά του κοσυφοπαίδιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Βέγγαλ. Δεν είναι παρόν. Ο κύριος Στογιάνοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα εναντίον της στρατηγικής διεύρυνσης γιατί έχει μια πολύ κολακευτική αντιμετώπιση της προόδου που έχει επιτύχει η Τουρκία σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλάβετε το μια και για πάντα η Τουρκία πριν από 100 χρόνια διέπραξε μια γενοκτονία εναντί άλλων εθνών. Σήμερα εξακολουθεί να διαπράττει γενοκτονίες. Η πολιτική της ελίτ χαίρεται για το γεγονός αυτό. Πριν από 20 χρόνια η Τουρκία υποστήριξε τρομοκρατικές οργανώσεις. Εξήγαγε την τρομοκρατία και εξακολουθεί να διατηρεί στενές σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος το οποίο είναι υπέρμαχος της τρομοκρατίας, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνώ. Ευχαριστώ κύριε Στοιόροφο. Κύριο Τάκουλα. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να φέρω στην επιφάνεια, αν θέλετε, ένα σημαντικό θέμα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης θα γίνουν σεβαστά. Και αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις χώρες οι οποίες θέλουν να, γίνει μέλη, να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας έκφρασης θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Σήμερα ψηφίσαμε και για τα δικαιώματα των γυναικών, θυμίζω. Θα πρέπει οι γυναίκες λοιπόν να έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς βία θα πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών να γίνονται σεβαστά σε όλες τις χώρες και υπογραμμίζομαι στην Τουρκία. Η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές και γρήγορες αλλαγές για να καταστεί έτοιμη να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γενιά μας δεν θα το γνωρίσει αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταίος και ίστατος ο κ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ ψήφισα όχι γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να τηρήσει όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης που θα του δώσουμε μια θετική γνώμη για αυτό το θέμα της ένταξης. Εξακολουθεί να υπάρχει μια συνοριακή διένεξη μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και δεν έχει ακόμα τελειώσει η παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους από την ε, Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τι άλλε χώρε, όμω τι χώρε των Βαλκανίων, θέλω να τι καλωσορίσουμε το ταχύτερο δυνατό εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κ. Κάτσμαρέκ για το, τη βία κατά των γυναικών. Πρόεδρε, δεν ε, στη συγκεκριμένη ψηφοφορία παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω γιατί τα θέματα της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μαζί από κοινού με τα θέματα αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Χτες, για παράδειγμα, κατηγορήθηκε η Καθολική Εκκλησία ως έναν από τους πιο βασικούς καταπιεστές των γυναικών. Αυτό είναι παράλογο. Στην Πολωνία δεν υπάρχουν επιλεκτικές αμβλώσεις, δεν υπάρχουν καταναγκαστικές ε, και Τέτοιε καταναγκαστικέ αιμομιξίες. Δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση των γυναικών σε ό,τι αφορά τον νόμο και δεν ε, καταδικάζονται όλες οι πράξεις βίας κατά των γυναικών από εκπροσώπους και των ε, δημοσίων αρχών αλλά και τη εκκλησία. Και γι' αυτό λοιπόν και αποκολούθησα την οδό τη εποχή. Ευχαριστώ. Ο επόμενος, ο συνάδελφο Μωτή. Signor εγώ υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος που καταδικάζει τη βία εις βάρος των γυναικών και αφιέρωσα την ψήφο μου στα 7 εκατομμύρια ταλίδων οι οποίες καθημερινά υφίστανται τη βία των ανδρών. Και φυσικά εκφράζω την αλληλεγγύη μου σε όλες τις γυναίκες της Ευρώπης. Προσπαθήσαμε να πιστέψουμε ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί στο εσωτερικό του πολιτισμού μας. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια ότι συμβαίνει μόνο στον οικιακό χώρο, αλλά γενικότερα και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Μην ξεχνάμε και τους ηλικιωμένου. Οι ηλικιωμένοι δεν υφίστανται μόνο φυσική βία, αλλά υφίστανται πολιτιστική βία, λέει ο όπως και τη στέρηση ελευθερίας κίνησης. Οι γυναίκες επίσης ε, υφίστανται τη βία αυτή και ε, σε πολύ μικρή ηλικία και αυτό χαρακτηρίζει φυσικά την περαιτέρω ζωή τους. Πρέπει να κάνουμε πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να μην μείνουμε σε επίπεδο καλών προθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Μότη. Εκ. Εκ. Εκ. Κυρία Ick. Ευχαριστώ κύριε Η βία κατά των γυναικών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η Σουηδία με 9 εκατομμύρια κατοίκου έχει 380 περιπτώσει βία κατά των γυναικών. Τώρα πέμπτο του γυναικείου πληθυσμού υφίσταται βία και ένα μεγάλο ποστόλο των γυναικών έχουν υποστεί βία σε κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό είναι πραγματικά ένα έσχο το να υπάρχει βία στον χώρο τον οικογενειακό που πλήττει την ακαιρεότητα των γυναικών αυτών. Οι γυναίκε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της ακαιρεότητα της προσωπικότητας του. Αυτή η μάστιγα σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι είναι απαραίτητο να αγωνιστούμε όλοι για την ισότητα των γυναικών. Έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραγνωρίσει αυτή την ζωφερή κατάσταση. Εγώ χαίρομαι για αυτό το ψήφισμα λοιπόν για την βία κατά των γυναικών και ζητώ από την ε, νέα Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της στο θέμα αυτό. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα μας υποβάλει νέες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Ευχαριστώ, κυρία Ικ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού με όλη μου την καρδιά, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας από όλο το πολιτικό φάσμα για να πετύχουμε ένα κοινό στόχο, να καταδικάσουμε και να καταργήσουμε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των γυναικών σε καταστάσεις συγκρούσεων στην Βοσνία Ζεγοβίνη, όπου έχω ζήσει την ε, κατάσταση και σε ό,τι αφορά τον Ταρφούρ επίσης. Νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια μας για να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σουηδική Προεδρία που συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θα αγωνιστώ για να καταστεί αυτό και προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματο τη Στοχόλμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Άλλο ένας ζητάει το λόγο για επεξήγηση ψήφου. Ο συνάδελφο σε αύριο, αλλά θα ήθελα να πω ότι τα αιτήματα για επεξήγηση ψήφου θα πρέπει να έχουν φτάσει στον Πρόεδρο πριν από την έναρξη. Κατ' εξαίρεση σας δίνω το λόγο. Στα υπόλοιπα θέματα όμως θα τηρήσω τη διαδικασία. Ο συνάδελφος της ΕΟΠΟ. Ah, Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. E, dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podkreślić, że temat Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα της βίας κατά των γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να επιληθεί του θέματο αυτού. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξή: ότι υπάρχουν βίες και ομέ πράξεις βίας σε βάρος των γυναικών, οι οποίε δυστυχώ σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε δεν έρχονται στην επιφάνεια και δεν την χάνουν της κατάλληλης απάντησης από τα δικαστήρια. Μερικές φορές οι ποινές είναι ιδιαίτερα επίηγείς. Αυτό το οποίο <clears throat> επομένως είναι ποινές οι οποίες είναι πραγματικά δυσανάλογα ελαφρές σε σχέση με τη βαρύτητα των ε, αδικοπραξιών κατά των γυναικών. Πολλές φορές λοιπόν γίνονται πράξεις οι οποίες μένουν ατιμόρυτες. Ουσιαστικά πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ιδίως αυτές οι οποίες είναι πράξεις βίας κατά των γυναικών. Μόνο με τις κατάλληλες τιμωρίες θα εξασφαλίσουμε ότι μια γυναίκα που είναι θύμα ενός τέτοιου αδικήματος μπορεί να τύχει ικανοποίησης από τα δικαστήρια. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα συναφή αδικήματα με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει τις επεξηγήσεις ψήφου για τη βία κατά των γυναικών. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της πειρατείας στην Σομαλία. Θέλετε διαδικαστική παρέμβαση. Επεξήγηση ψήφου για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Συνάδελφε, ο κανονισμός προβλέπει το εξή. Θα πρέπει να ολοκληρώνουμε το ένα θέμα μετά το άλλο και έχουμε είχαμε φτάσει στο θέμα της εξάλληψης της βίας εναντίον των γυναικών. Τώρα περνάμε στο θέμα της πολιτικής λύσης για την πειρατεία στη Σομαλία. Όλα με τη σειρά τους και για την επεξήγηση ψήφου, αυτά, έχουμε, ε, ψήφου αυτή έχουμε τον κύριο Μπούντες. Πρόεδρε, το κόμμα για την ελευθερία ψήφισε κατά της ψηφίσματος αυτού και να εξηγήσω γιατί. Θεωρούμε ότι η παρακολούθηση των πλοίων αποτελεί καθήκον του ΝΑΤΟ. Δεν έχει στρατό η Ευρώπη και δεν έχει να κάνει τίποτα εκεί. Είναι 100% καθήκον του ΝΑΤΟ. Επίσης, το κόμμα της Ελευθερίας πιστεύει ότι τα πλοία εμπορικής ναυτιλίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν σε αυτές τις επιθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να τεθεί ένα τέρμα στην πειρατεία στη Σομαλία, όχι όμως με τον τρόπο αυτό. Ähm, Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπόντες, ήταν μοναδική επεξήγηση ψήφου για το συγκεκριμένο θέμα και περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος για το περιβάλλον χωρίς καπνό. Η συνάδελφος Ζαμπόσκα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συστάσεις για τον χώρο κατά, χωρίς ε, κάπνισμα έχουν σε στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να προστατευτούν από το παθητικό κάπνισμα σύμφωνα με το πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνίσματος. Τονίζω ότι το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι η πιο συχνή αιτία για θανάσιμες ασθένειες όπως είναι καρδιοαγιακά προβλήματα, ε, καρκίνος των πνευμόνων κτλ. Υπάρχει και θέμα μείωσης της γονιμότητας των νέων ανδρών και γυναικών που δεν αναφέρεται τόσο συχνά. Επίσης, ό,τι αφορά τη δημογραφική κρίση και ενώ αναπτύσσουμε νέες τεχνητές μεθόδους γονιμοποίησης, θα έπρεπε παράλληλα να αυξήσουμε και τη συνειδητοποίηση για τις οικογένειες να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις αρνητικές συνέπειες του καπνού τις είναι συνέπειες του καπνού και επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια παρακολούθηση και της δράσης της βιομηχανίας ε, τσιγάρου για να μην υπονομεύσουν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω δύο πτυχές σε ό,τι αφορά τα περιβάλλοντα χωρίς καπνό. Καταρχάς ε, ψήφισα υπέρ ε, της αρμοδιότητας των κρατών μελών για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί θεωρώ ότι σωστό είναι να λέμε ότι καταρχάς έχουμε την αρχή της επικουρικότητας, αλλά δεν έχουμε λοιπόν και αρμοδιότητα, αλλά από την άλλη είμαι υπέρ του περιβάλλοντος ε, χωρίς καπνό και θα πρέπει να τηρήσουμε τις ισορροπίες. Μια δεύτερη πτυχή είναι ότι πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία επιδοτεί την καπνοπαραγωγή και γι' αυτό λοιπόν ψήφισα όπως ψήφισα, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό συνάδει με την προσπάθεια καταπολέμησης και μείωσης του καπνίσματος. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να επιτύξουμε συνέπεια. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον καπνό, να μην επιδοτούμε και την καπνοπαραγωγή. Κυρία ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι. Η ομάδα της Τσέσου θέλει να έχει σαφείς και εφικτού και εφαρμόσιμους κανόνες που να ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ευρώπη αλλά όχι κανόνες οι οποίοι να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλές χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κανόνες και σε άλλες επίκειται η εφαρμογή τέτοιων κανόνων. Εγώ δεν πιστεύω, όπως η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται να πιστεύει, ότι όλοι οι κανόνες για την προστασία των, από το παθητικό κάψιμα πρέπει να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Υπάρχει αρμοδιότητα μονάχα σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων και για μένα αυτό είναι πρόβλημα, γιατί είναι πιο σημαντική η προστασία των παιδιών και των νέων. Αυτή είναι μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες και δεν έχει νόημα να έχουμε κανόνες οι οποίοι περιορίζονται μονάχα στον τομέα τη εργασία και δεν λαμβάνουν υπόψη την προστασία των νέων και των παιδιών. Εγώ επομένω υποστήριξα την τροπολογία αυτή που επισημαίνει αυτό το γεγονό και χαίρομαι που ενεκρίθη αυτή η τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Γκέ Βάι Γκέρμπερ. Η κυρία Χάρκιν τώρα έχει το λόγο. Προέρχομαι από μια χώρα όπου έχουμε απαγορεύσει το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους εδώ και καιρό και ήμουν μέλος της Ιρλανδικής Βουλής τότε και υποστήριξα την απαγόρευση. Έχουμε διαφορετικές απόψεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. Και υπάρχει θέμα σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, υπάρχει νομοθετική αρμοδιότητα εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεσή του σαν παράδειγμα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά στις χώρες όπου υπάρχει η απαγόρευση του καπνίσματος δεν θα πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας στον τομέα της εστίασης. Μιλήσαμε χθε για τις εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων στους τομείς της επικουρικότητας στα πλαίσια της νέας συνθήκης. Πρέπει να είμαστε πολύ συνεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε από εδώ και πέρα. Συζητούσαμε συναδέλφους ε, στην αρχή και έχασα την ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση του Κοινοβουλίου και ήμουν από τις πρωταγωνίστριες στο προηγούμενο κοινοβούλιο που όρισαν το 11 σαν χρονιά του εθελοντισμού. Ο κύριος Γκόλνης. Κύριε Πρόεδρε, είμαι λίγο συγκινημένος γιατί η μητέρα μου γεννήθηκε στην καπνοβιομηχανία του Στρασβούργου όπου εργαζόταν και ο παππούς μου που μόλις έκλεισε το εργοστάσιο αυτό. Τότε ήταν δημόσιο το εργοστάσιο, έγινε ανώνυμη εταιρεία, ιδιωτικοποιήθηκε και είχαμε εξηγήσει στους εργαζομένους ότι δεν υπήρχαν συνέπειες στην απασχόληση. Ανησυχεί ο κόσμος, ανησυχούν και άλλοι κλάδοι του δημοσίου που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες απειλές. Κατανοώ βέβαια και νομιμοποιώ την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού, προϊόντων καπνού. Αλλά δυστυχώς η γαλλική παραγωγή έχει εξαφανιστεί η κατανάλωση του Στρασβούργου έκλεισε, αλλά παρόλα αυτά η κατανάλωση του τσιγάρου συνεχίζεται με καπνά τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ ναι μεν υποστηρίζω την τιμή η οποία δίδεται για τους καπνοκαλλιεργητές εφόσον καταναλώνεται καπνό στην Ευρώπη καλύτερα να παράγεται εδώ παρά να εισάγεται από αλλού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Υποστηρίζω απόλυτα όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον αγώνα για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Αλλά αυτές οι δράσεις δεν θα έπρεπε να εστιάζουν στο να περιορίσουν την επιδότηση για την καλλιέργεια καπνού. Γιατί η καπνοπαραγωγή δεν έχει άμεση σχέση με την κατανάλωση του καπνού. Αν περιορίσουμε ή αν εξαλείψουμε την παραγωγή καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αντίστοιχους αγρότες, <clears throat> θα παραμείνει η κατανάλωση εισαγόμενου καπνού και καπνικών προϊόντων. Δεν είναι ο τρόπος λοιπόν με αυτός με τον οποίο θα μειώσουμε την κατανάλωση του καπνού στην Ευρώπη. Είναι σαν να προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση πύρας μεταξύ των νέων με το να, με αγωνιζόμαστε εναντίον των ζηθοποιείων. Επομένως υποστήριξα όλους αυτούς που είπαν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης καπνού. Ευχαριστούμε. Έχουμε τελειώσει και με αυτό το ψήφισμα και ερχόμαστε στο τελευταίο ψήφισμα που είναι <clears throat> επιστηστική ασφάλεια διάσκεψη κορυφής του ΦΑΟ. Η κυρία Σαμπόσκα έχει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η επιστηστική κρίση δεν αποτελεί μόνο θέμα επιστηστικό ή οικονομικό. Επηρεάζει και την ε, παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη. Υποστηρίζω ότι υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στο ψήφισμα, γιατί δεν κινηθήκαμε προς την, κατάστα... προς την κατεύθυνση που θέλαμε, παρά το γεγονός ότι η πείνα αποτελεί ένα φαινόμενο με πολλαπλές διαστάσεις. Η συζήτηση περιορίστηκε στα τεχνικά στοιχεία. Και ο κύριος Ζάκοντιφ απογοητεύτηκε και από τη συζήτηση αλλά και από το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των δυτικών χωρών δεν συμμετείχαν και ε, από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θεωρώ ότι η πείνα και η φτώχεια αποτελεί ένα θέμα για τα μέσα μαζική ενημέρωση τελικά για τον τύπο και όχι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί κατεπηγόντω. Κάποιο θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε αυτέ για του ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ, συνάδελφε, και ήταν και τελευταία επεξήγηση ψήφου. Γι' αυτό διακόπτουμε μέχρι τις 3.